ειδικά εσείς που βρίσκεστε εδώ για τελευταία φορά. Η συμφωνία αυτή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστερημένου στο πολιτικού ρεαλισμού. Το σημερινό ψήφισμα το δέχεται. Πρέπει όμως να αναφέρουμε τρία σημεία. Πρώτον, η συμφωνία ορίζει ότι στο μέλλον ε, τα μέρη μπορεί να δέχονται ταυτότητες χωρίς έλεγχο βιομετρικών στοιχείων. Κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο προφανής οικονομικός λόγος ή νομικός ή λόγος ασφαλείας. Ε, βεβαίως έχουν τεθεί ζητήματα ιδιωτικότητα. Ε, κάτι το οποίο ξεχνάμε παρά το ότι συνεχώς αγωνιούμε υποτίθεται για τα δικαιώματα. Δεύτερον, η συμφωνία παγώνει τα δικαιώματα όπως αυτά ερμηνεύονται σήμερα, ενώ η μελλοντική ερμηνεία παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ένωσης. Ουσιαστικά ζητείται εδώ πέρα από το Δικαστήριο να διαμορφώσει δύο νομολογίες. Μία για τα δικαιώματα των υπηκών των 27 και μια άλλη νομολογία για τη Βρετανία με βάση το δίκαιο προ-Brexit. Πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ε, Το άρθρο 18 του ψηφίσματος εκφράζει την λύπη του για το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τερματίσει την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων και λέει ότι οι τέσσερις ελευθερίες είναι αλληλένδετες και οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να είναι υπό την αίρεση του να δεχθεί την ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων το Ηνωμένο Βασίλειο. Το αίτημα αυτό στρέφεται κατά των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης. Οι συμφωνίε ελευθερίου εμπορίου, οι περισσότερε μάλιστα τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κανόνα δεν λένε τίποτα για την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων. Το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εμπορικό πλεόνασμα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε είναι προ το συμφέρον τη Ένωση να έχουμε μία συνολική εμπορική συμφωνία. Αν μιλάμε σοβαρά για τα δικαιώματα των πολιτών, τότε οι πολίτες της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να έχουν και τα οικονομικά τους συμφέροντα τα οποία θα γίνουν σέβαστα. Σας ευχαριστώ. Φαν για το ECR για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πως η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν Είχε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον ε, Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πήγαν πολύ καλά, θετική ατμόσφαιρα, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Τώρα πρέπει να σημειωθεί γρήγορη πρόοδος για την ε, μελλοντική μας ε, σχέση. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκρίνουμε τη συμφωνία. Όπως ξέρετε η Βουλή των Κοινοτήτων την ενέκρινε με μια πλειοψηφία 99 ψήφων Τώρα έχει πάει στην Βουλή των Λόρδων και πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την συμφωνία αυτή για να τεθεί ενισχύ στις 31 Ιανουαρίου. Και φαντάζομαι θα γίνει αυτό ομαλά. Βεβαίω ο έλεγχο των ε, συνόρων μα ήταν ένα σημαντικό ε, παράγοντα στην απόφαση αποχώρηση. Πρέπει να το έχει κατά νου αυτό η κυρία Χούμπνερ. Για τα δικαιώματα των πολιτών. Εδώ και η Βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πολύ συμφωνούν. Μου αρέσει η πρώτη παράγραφος εδώ πέρα, λέει θεωρεί ότι το μέρος δεύτερο είναι δίκαιο και ισορροπημένο. Εκεί πρέπει να σταματάει το ψήφισμα ουσιαστικά. Βεβαίω, εντάξει, να βοηθήσει θέλει το ψήφισμα παρά τι παρεξηγήσει και κάποιε γκρίνιε. Το ελπίζω, αλλά ελπίζω να βρεθεί και κάποιος ρόλος για τον κύριο Φερχόφστατ στο μέλλον. Ιστορικά βεβαίως καμία χώρα δεν ε, προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου περισσότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το ψήφισμα εστιάζει δυσανάλογα στο μελλοντικό καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών στην Ένωση, ενώ δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου με τους Βρετανούς πολίτες στις 27 χώρες. Μία παράγραφος από τις 22. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο των ετοιμασιών, αλλά τα κράτη-μέλη δεν έχουν σχέδια για το πώς θα λειτουργεί το σύστημα για τους Βρετανούς πολίτες. Όπως και οι Βρετανικές αρχές θα φροντίσουν όσους κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω στο μέλλον, απουσία Ευρωπαίων Ευρωβουλευτών, το Κοινοβούλιο αυτό μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια να φροντίσει να διασφαλίσει τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ΚΟΕ Σύρδευαν. δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε για τα δικαιώματα αυτών που συνεισφέρουν στην ευημερία της ε, Βρετανικής κοινωνίας, είτε στην οσυλία, είτε στην έρευνα, είτε ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίε. Βεβαίω δεν θα κλείσουμε τον δρόμο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολίτες Βρετανοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, έχουν τα δικαιώματα τα οποία είχαν. Βεβαίως η συζήτηση αυτή είναι σημαντική γιατί υπάρχει ανησυχία ε, για τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία θα μπορούσαν να πληγούν στην διαδικασία αποχώρησης. Αυτό αφορά κυρίως την άδεια παραμονής, ε, αλλά και το πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες αυτές για ευπαθή άτομα ηλικιωμένους. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τις ε, περαιτέρω σχέσεις μας, οι οποίες είναι πολύ ευρύτερες ε, από εμπορικές σχέσεις, αφορούν ε, οικονομικές, οικολογικές ε, σχέσεις, όλα αυτά θα μας απασχολήσουν και στις δύο χθες της μάχης και δεδομένων των πολιτικών πτυχών είναι νομίζω ε, σαφές ότι δεν μιλάμε για μια απλή εμπορική συμφωνία που μπορεί να ολοκληρωθεί σε 11 μήνες. Δηλαδή μην ε, έθελο τυφλούπε. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Μπόρις Τζόνσον, η κυβέρνησή του, θα πρέπει να ζητήσει εγκαίρως μια παράταση για να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών, έτσι ώστε να έχουμε όλοι τον χρόνο που χρειαζόμαστε. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Αν δεν γίνει αυτό, το τονίζω αυτό, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit με όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει αυτό. Η ομάδα μου τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπέρ Διασφάλιση τη ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό θα το κάνουμε και στο μέλλον. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει πτώση των προδιαγραφών γιατί θα έχει την ιδέα η Βρετανική κυβέρνηση πως θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω dumping. Αυτό δεν πρέπει να γίνει ούτε σε φορολογική πολιτική, ούτε στα κοινωνικά, ούτε σε οικολογικά ζητήματα, ούτε στην προστασία των καταναλωτών. Και τέλος, ε, δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τους Βρετανούς εκείνους συναδέλφους με τους οποίους είχαμε μια επικοδομητική συνεργασία για μια καλύτερη Ευρώπη. Θα μας λείψατε. Ευχαριστούμε. Από τους μη εγγεγραμμένους, ε, κυρία Φιλίπς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεκινήσει την ε, συζήτηση και ε, το πρόγραμμα αυτό. 13 χρόνια τα συζητάμε. Ότι όσοι έχουν ε, κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο σπίτι του θα πρέπει να παραμείνουν με ίδιου όρου και δικαιώματα με όλου του υπόλοιπου. Αλλά όχι περισσότερα δικαιώματα για εκείνου. Δεν θέλουμε ευνοιοκρατία εδώ πέρα, γιατί εσείς ουσιαστικά προτείνετε ε, οι Αφρικανοί, οι Ασιάτες, οι Αμερικανοί και όλοι οι υπόλοιποι που επίσης έχουν έρθει να μείνουν στον Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το σπίτι τους κάπως ε, είναι σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και εμείς δεν συμφωνούμε αυτό, δεν είναι ε, αυτό αξία του έθνους μου. Ακούω υποτίθεται έναν επικοδηματικό διάλογο σήμερα, αλλά Προτείνω σε όλους αυτούς που ακολουθούν την ε, τρομολαγνία ε, τελευταία να τους υπενθυμίσω ότι το Νέο Βασίλειο είναι μια ανοιχτή και φιλόξενη χώρα. Μην ε, σπέρνετε λοιπόν τον τρόμο στον κόσμο. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού γιατί θα γίνουμε ανεξάρτητο έθνος με ανεξάρτητη μεταναστευτική πολιτική και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να προστατεύονται όλοι. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκονσάλες Πόνς για ένα μισή λεπτό. Να μιλήσω αγγλικά γιατί θέλω να ακουστώ στα αγγλικά. Ο Βρετανικός λαός θα πρέπει να ξέρει ότι παρά το Brexit και παρά όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία τέσσερα έτη πάντοτε θα είναι ευπρόσδεκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Ευρώπη δεν έχει να κάνει με το που προέρχεσαι αλλά το που θες να πας. Οι χώρες ε, μπορεί να χωριστούν αλλά οι οικογένειες όχι. Σήμερα έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο Βρετανούς που ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πολλοί και στην Ισπανία, στη χώρα μου. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτού σήμερα απευθεία. Πολλοί από εσά έχετε φτιάξει τη ζωή σα εδώ στην Ευρώπη. Πολλοί από εσά έχετε παντρευτεί εδώ και κάποιοι έχετε παιδιά που γεννήθηκαν εδώ. Είμαστε γείτονες και πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι και συγγενείς υπάρχει κάτι που δεν θα ξεχάσουμε, ούτε μπορούμε να το ξεχάσουμε. Γι' αυτό θέλω να σας πω, ό,τι και να συμβεί μετά την 31η Ιανουαρίου, εσείς πάντοτε θα νικείτε στην Ευρώπη. Και όσο είναι η ιανουαριου εσεις παντοτε θα νικετε στην ευρωπη και οσο ειναι η επιθυμια σας να μείνετε μαζί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε θα είναι το σπίτι σας. Επομένως, από τα βάθη της ψυχής μου, δεν θα πω ε, αντίο, δεν θα πω στο επανειδήν, θα πω μόνο μείνετε μαζί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και το δικό σας σπίτι. Ευχαριστώ. πολύ. Για ένα λεπτό, κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στην ε, Επιτροπή Αναφορών ακούσαμε πολίτες από όλη την Ευρώπη που με απελπισία σκέφτονται τι θα γίνουν τα δικαιώματά τους, οι ζωές τους, οι δουλειές τους, οι οικογένειές τους. Όταν ε, τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία, ε, μάλλον ανησυχούν αυτοί οι άνθρωποι για το τι θα γίνει μετά την μεταβατική περίοδο. Γιατί όλοι αυτοί δεν είχαν καμία φωνή στην απόφαση που τελικά επηρέασε τόσο καθοριστικά τη ζωή τους. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν τις αξίες ε, των ε, ε, ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πάνω απ' όλα ένα ηθικό καθήκον προς εκείνους που δεν κατάφεραν, δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν και δηλώνουν την απογοητευσή τους. Συνεχώς δηλώνουμε ότι η διασφάλιση των, των δικαιωμάτων των πολιτών είναι κόκκινη γραμμή για οποιαδήποτε συμφωνία για τον Brexit. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε και να εμείνουμε σε αυτή τη θέση. Πρέπει να επιδείξουμε θάρρος, και να ζητήσουμε περισσότερε ενέργειε πριν ψηφίσουμε επί τη συμφωνία αυτή την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, κυρία Βόνταν, για ένα λεπτό. Emmanuel Είναι δασκάλα η Εμμανουέλ και έχει διδάξει χιλιάδες εφήβους ε, στα βρετανικά σχολεία, έχει πληρώσει τους φόρους της, έχει παντρευτεί Βρετανό και έχει παιδιά που είναι Βρετανοί. Πρόσφατα ε, ζήτησε το καθεστώς ε, εγκατάστασης και επέλεξε να γίνει πατρίδα της χώρα όπου έχει δουλέψει, πληρώσει τους φόρους και εργαστεί στην κοινότητα της. Και αρχικά της αρνήθηκαν αυτό το καθεστώς εγκατάστασης. Στο να διασφαλίσουμε ε, τον, τα δικαιώματα των τριών εκατομμυρίων πολιτών που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι θεμελιώδε. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά του να αποκαλούν το Ηνωμένο Βασίλειο την πατρίδα του. Πρέπει να υπάρχει αμοιβή αναγνώριση προσωπικών επαγγελματικών προσόντων. Δεν υπάρχει κανένα ε, λογικό λόγο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια αναγνωριστική διαδικασία η Βρετανική κυβέρνηση για να δώσει το καθεστώ με ένα υλικό έγγραφο και να συνεχίσει την ανεξάρτητη παρακολούθηση αυτή τη διαδικασία. Αν αποτύχει να το κάνει αυτό, δυστυχώ ντροπιάζει η κυβέρνηση τη χώρα μα και θέλω να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη επίση να ανταμείψουν με τον ίδιο τρόπο ε, του Βρετανού πολίτε που ζουν στα κράτη-μέλη. Αν θέλετε, κύριε Τζόνσον, να έχετε μια καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που να λειτουργεί, γιατί δεν ξεκινάτε σεβόμενο τα δικαιώματα τριών εκατομμυρίων και αποφεύγοντα τη δυνατότητα να έχουμε ε, και πάλι μια χαμένη γενιά. Κύριε Βανόρντεν, θέλει να σας θέσει μια ερώτηση, κύριε Βόντεν. Δέχεστε. Η απάντηση είναι όχι. Για ένα λεπτό, ο κύριος Σαλάρ. Ευχαριστώ. Είμαι ένας από τους ε, επικόους Ευρωπαϊκής Ένωσης που του ζήτησαν να ε, ζητήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα κατάστασης. Πάνω από 35 χρόνια ζω στη Σκωτία ε, και πήγα λόγω της ελευθερίας μετακίνησης. Δεν καταλαβαίνω πώς καταλήξαμε εκεί. Το, το σύστημα αυτό του Ευρωπαίου, του, της Βρετανίας δεν είναι κατάλληλο. Πώς ε, ε, μπορεί να προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του υπηκόου που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το θέμα ήταν ένα από τι κόκκινε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ποιο τη συμφωνία, θέλω να σα επενθυμίσω. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικά θα είναι το τελευταίο που θα αποφασίσει επί της νομοθεσίας. Ε, όμως ε, πόσο αξίζουν ε, όλα αυτά, αυτό το έγγραφο, πόσο αξίζει η εμλήξη μετά από 8 έτη και είδαμε τι συνέβη με το δικαστήριο αυτήν την εβδομάδα. Εγώ έχω αμφιβολίες και ανησυχώ πάρα πολύ για το τι θα συμβεί στο μέλλον το πρόγραμμα κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι κατάλληλο. Εγώ δεν θα ζητήσω να ενταχθώ για να μου το δικαίωμά μου να ζω ε, στο σπίτι μου. Η διαδικασία της αίτηση ε, θα πρέπει να καταργηθεί. Τα δικαιώματά μα θα πρέπει να προστατεύονται αυτόματα. Και οι άνθρωποι που ζουν ε, στη Σκωτία θεωρούν ότι η Σκωτία πρέπει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, βέβαια, στο επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Ελάρτ, ο κύριος Βανόρντερ θα προσπαθήσει εκ νέου να θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε. Δέχεστε την ερώτηση από τον κύριο Ορντερ. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρο στα γαλλικά. Αν, αρνηθείτε, αν σας αρνηθούν και τρίτη φορά, θα τα εγκαταλείψω. Να δούμε τι θα γίνει όμω. Λοιπόν, είμαι σε καλή διάθεση για να ακούσουμε αυτό το ενημερωτικό θέμα. Σας ευχαριστώ για την ενοχή σας, Πρόεδρε στους δύο τελευταίους συνάδελφους που μίλησαν. Θέλω να πω. Έχουμε 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μόνο σε πέντε ε, τους αρνήθηκαν ε, λόγω ποινικού δικαίου. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Βερνόρντεν. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Δεν ε, ήταν ερώτηση, ήταν διαδικαστικό και θα σας επιτρέψω για 30 δευτερόλεπτα θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το διαδικαστικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω. Γιατί και το, το έχουμε ξανακούσει αυτό ότι οι περισσότεροι που έκαναν έτσι κατάφεραν να λάβουν το καθεστώς. Όμως ε, το 47% των ετούντων έτυχαν απόρριψης και πρέπει να ξανακάνουν αίτηση. Αν κάνεις αίτηση και σου αρνούνται και φυσικά σου αρνούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι απορρίφθηκαν ε, και πηγαίνετε πίσω στο Λονδίνο να τα πείτε στον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Βανόρντεν, όχι. Εγώ ήμουν πρόθυμη να το λόγο, αλλά όχι τώρα. Ο κύριος Τέρτς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με το Brexit η αλήθεια είναι ότι ε, πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανοχή και αν είχαμε κάτι τέτοιο ίσω θα είχαν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Βρετανοί γιατί ε, ίσως τέτοιες συμπεριφορές εξηγούν πολλά. Με το Brexit στι 31 Ιανουαρίου υλοποιείται η βούληση του Βρετανικού λαού. Αυτή η απόφαση των Βρετανών θα έπρεπε να έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτοκριτική. Όμω το αντίθετο έγινε. Αντίθετη η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέθηκε σε όποιον αποχωρεί. Εμεί λυπούμαστε για το Brexit. Οι Βρετανοί έχουν δύο μεγαλέ αρετέ. Ε, το θάρρο και την αγάπη προς την ελευθερία. Τους χρειαζόμαστε εδώ από μέσα εμείς που αντιμετωπίζουμε τις ηγεμονικές ιδεολογικές τάσεις και τα φεντερελιστικά όνειρα κατά των εθνών. Στην Ισπανία ζουν 250.000 Βρετανοί, στο Ηνωμένο Βασίλειο 180.000 Ισπανοί τα δικαιώματα και των μεν και το δε θα πρέπει ε, να τα εγγυηθούμε εξίσου. Γι' αυτό έχουμε πολλούς λόγους ε, να ε, έχουμε αμοιβαιότητα. Οι σχέσεις με το Λονδίνο φαίνεται να είναι πιο εύκολες από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παρά από τις Βρυξέλλες, γιατί από τις Βρυξέλλες φαίνεται να υπάρχει ένα πνεύμα ρευαρσισμού που θα κάνει όλα πιο δύσκολα. Η κυρία Ρέγο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι στις 31 Ιανουαρίου θα έχουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω σεβόμαστε τη δημοκρατική απόφαση του Βρετανικού λαού από την Ισπανία. Πιστεύουμε όμως υπήρχαν κάποιοι άγνωστοι παράγοντε που θέλουμε ε, να προσεγγίσουμε. Είναι ιδιαιτερότητα η περίπτωση του Γιβραλτάρ. Μιλάμε για ε, πάνω από 13.000 ε, εργαζομένους που κάθε μέρα περνούν τα σύνορα. Και είχαμε στην περίπτωση του Γιβραλτάρ, ε, μεταμόρφωση μία ε, από τι πιο φτωχέ περιοχέ τη Ευρώπη. Έχουμε 27% ανεργία και στου πιο νέου 70%. Ακόμη και αν το άρθρο 24 Συμφωνία Αποχώρηση ε, υποθέτει ότι υπάρχει μία πρόοδο τη κατάσταση, δεν λαμβάνει κανένα μέτρο που να εγγυάται ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν δικαιώματα όπω επιδόματα ανεργία ή τη σύνταξή του. Με τη συμφωνία αυτή εγγυώνται τα δικαιώματα των οικονομικών ελλήνων είναι Εμείς τώρα ζητάμε την απόλυτη δέσμευσή τους έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην μείνουν εκτός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Βούντικομ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα παρακαλώ να επικεντρωθώ στην παράγραφο 18 του εγγράφου που αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο με τα διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι θα τεθεί τέλος ε, στην ελεύθερη μετακίνηση. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι το τέλος της ελεύθερης μετακίνησης ήταν ένας ε, ε, κύριος παράγοντας σε ό,τι αφορά την απόφαση του Βρετανικού λαού να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πραγματικά μία κινητήριος δύναμη αυτής της απόφασης. Και όμως βλέπουμε εδώ σήμερα ότι υπάρχει μια πολιτική δισκαμψία και μοιοπίας προς αυτό. Δεν θέλετε να το δείτε. Τώρα λέτε για την ε, διαδικασία αίτησης. Δεν πρέπει καν κανείς να τολμήσει να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για να ε, στοιχειοθετήσει με τέτοια αίτηση. Οι Βρετανοί πικοί ζητούν από την ε, Βρετανική κυβέρνηση να δώσει τέλος στην ελεύθερη μετακίνηση και με αποτελεσματικό μάλιστα τρόπο, όχι μόνο ε, κατόνομα. Και πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καταλάβει για να κάνουμε επιτέλους μια σωστή συζήτηση. Κυρία Βιντεκόμ, η κυρία Νιτφέλτ θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Το δέχεστε? Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βιντεκόμ, άκουσα που είπατε ο Βρετανικός λαός θέλει το ένα και το άλλο. Όμω, δεν ισχύει ότι μόλις 43% ε, των πολιτών υπερψήφισε το δικό σας πολιτικό θεματολόγιο και μόνο και εξαιτία του Βρετανικού εκλογικού συστήματος κατάφερε ο κύριος Τζόνσον να πάρει την πλειοψηφία και στην ουσία η πλειοψηφία του Βρετανικού λαού δεν ψήφισε για τον Brexit, έτσι δεν είναι. 17,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην μεγαλύτερη ε, συμμετοχή σε δημοκρατικές εκλογές στη βρετανική ιστορία ψήφισαν την αποχώρηση. Εμείς ε, είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα σε αυτό το κοινοβούλιο. Γιατί γιατί ο Τζόνσον πήρε τέτοια ε, μαζική πλειοψηφία σε εκλογές, γιατί το βασική του δέσμευση ήταν να υλοποιήσει το Brexit. Mr. Rangel. Κύριε Ραντζέλ, έχετε το λόγο για ένα μισή λεπτό. Quiet, please. Could I ask our British colleagues to my right to be quiet, please? There's a speaker to take the floor. Παρακαλώ, κάτι ησυχία. Ο κύριος Ραντζέλ. Στο Συμβούλιο και η Επιτροπή και συγκεκριμένα στον κύριο Μπαρνιέ θέλω να πω τα εξής. Η Πορτογαλία που την εκπροσωπώ εγώ, είναι μια χώρα που έχει την ε, πιο παλιά συμμαχία του κόσμου με το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1386 και ε, αναφέρθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και ε, ισχύει. Λίγες ε, χώρες ε, θα λυπηθούν ε, τόσο πολύ για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου όπως εμείς, όμως λίγοι θα δηλώσουν ότι θέλουν να έχουμε τους πιο δυνατούς συνδέσμους μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική η κατάσταση των πολιτών για μας και πολλά πρέπει να γίνουν και θέλω εδώ να σκίσω κριτική στη Βρετανική κυβέρνηση γιατί μερικές φορές φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί περισσότερο για την κατάσταση των Βρετανών ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την ίδια Βρετανική κυβέρνηση. Και γι' αυτό θέλω να απευθύνω έκκληση στην κυβέρνηση Τζόνσον, προκειμένου γρήγορα να θέσει σε εφαρμογή όλε τι διατάξει, οι οποίε έχουμε συμφωνήσει, έτσι ώστε οι πολίτε ε, και από τι δύο πλευρέ τη μάχη να μπορούν ε, να ζήσουν στα πλαίσια μια συνεργασία και μια φιλική σχέση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράης για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Μισελ Μπαρνιέ και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά σε αυτό το θέμα. Είναι η κοινή μας ευθύνη. Εμείς βρισκόμαστε εδώ γιατί το ψήφισμα αυτό αποτελεί προειδοποιητική βολή, παραπάνω από μία βολές, και ο κόσμος ανησυχεί. Γι' αυτό ακριβώς ε, είπαμε να ακούσουμε τι ανησυχίε ε, των ανθρώπων για τα δικαιώματα των πολιτών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργό προσφάτως στην απόφασή του να αναθεωρήσει το σχετικό νομοθέτημα για να επιτρέψει για να υπάρξει μια ανεξάρτητη αρχή γιατί υπήρξε ένα σχετικό σκάνδαλο με πολίτες από την Καραβική παλαιότερα ε, αποφάσισε να ενισχύσει την ανεξάρτητη αυτή αρχή. Δεδομένης της ιστορίας ε, των μεταναστευτικών αρχών, αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πηγαίναμε. Οπότε ας είμαστε σαφείς. Είναι σοβαρές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και έχουμε σοβαρές ανησυχίες για τους Βρετανούς πολίτες. Αν δεν τα καταφέρουμε θα έχουμε μια πληγή και μια αδικία η οποία θα, καθορίσει τις μελλοντικέ ε, συμφωνίες για πολλά χρόνια. Οπότε όταν μιλάμε για χάρτινο έγγραφο ή για ένα σύστημα δήλωσης, αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αδικίες που θα συνεχιστούν χρόνια χωρίς να υπάρχει κάποιος μηχανισμός επίλυσης και θα αποτελέσουν τμήμα της νομολογίας και του αφηγήματο. Γι' αυτό ο κύριος Μπαρνιέ θεώρησε τόσο σημαντικά τα δικαιώματα των ε, πολιτών ε, και γι' αυτό ακριβώς το ψήφισμα αυτό αποτελεί προειδοποιητική βολή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντουρόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δύο λόγια για να πω ποιο είναι ο λόγος που αυτό το ψήφισμα είναι τόσο σημαντικό. Είχα την εντύπωση, όπως και πολλοί συνάδελφοι, πριν ε, την παρέμβαση αυτή σήμερα, πως το θέμα των πολιτών ε, έπρεπε να είναι προτεραιότητα και στην καρδιά των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Και ήθελα ο κύριος Μισελ Μπαρνιέ, ξέρω ότι έχει συνείδηση αυτού, ότι το, το Κοινοβούλιο θα το υποστηρίξει ομόφωνα για να ε, υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει πιθανή συμφωνία αν δεν εντάξουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Είμαι πολύ πεπισμένο για αυτό που λέω τώρα και για την αναγκαιότητα του ψηφίσματο και για την αναγκαιότητα να το εγκρίνουμε ευρέω. Ε, ε η Βρετανική ακροδεξιά να έρχεται εδώ μετά από αυτά τα ψέματα και να έρχονται ε, να ζητάνε μία εμπορική συμφωνία χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων πολιτών είναι ντροπιαστικό και το δηλώνω μπροστά του. Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία αν δεν σεβαστείτε τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ένας κανόνας που θα σας επιβάλλει αυτό το κοινοβούλιο, είτε το θέλετε είτε όχι. Συνάδελφοι, έχουμε 16 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο στο KTI. Θα κλείσει εδώ ο κατάλογος. Περνάμε τώρα στην κυρία Ράιντ και για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. η ομιλία αυτή μάλλον θα είναι η δυσκολότερη που θα βγάλω. Εγώ κατέβηκα ω Ευρωβουλευτή για να παλέψω για περισσότερα δικαιώματα και τώρα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε θα χάσουν δικαιώματα και δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να το δω θετικά. Τέλος πλησιάζουμε το Brexit. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο θετικά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι απόλυτο σίγουροι για το ότι υπάρχουν Εκατοντάδε ευρωβουλευτέ που εργάζονται εδώ για να παραμείνει αυτό το κοινοβούλιο και δικό σα θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά σας εδώ. Δεύτερον, και απευθύνομαι στους Βρετανούς, ε, στους ανθρώπους του ΕΒ που αυτή τη στιγμή είναι απαρηγόρητοι. Ακόμα και με αυτό το κίνημα, το μοναδικό στην ευρωπαϊκή ιστορία, δεν καταφέραμε να έχουμε δεύτερο δημοψήφισμα. Όλες οι διαδηλώσεις αυτές ε, δεν ήταν μάτες, ε, φτιάξατε κάτι το υπέροχο τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο φιλοευρωπαϊκό κίνημα πολιτών που έχουμε δει και θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό και πιστέψτε με, μία μέρα θα επανέλθουν Βρετανοί Ευρωβουλευτές σε αυτή την αίθουσα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιντάντσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καθώς ε, ακούμε τους κύριους σχολιαστές, ε, λέγεται ότι ο Βρετανικός λαός εξέφρασε τη βούλησή του. Είτε μας όχι, αυτό αποκαλείται δημοκρατία. Τώρα όλοι καλούμαστε να οικοδομήσουμε μια νέα θετική συνεργασία μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών είναι μία από τις πιο ευαίσθητες στοιχές. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι γίνονται θετικά βήματα, ακόμη και αν πρέπει να βελτιωθούν σίγουρα οι γραφειοτικές διαδικασίες ε, για ε, να μπορέσουν ε, όσοι έχουν δικαίωμα να κάνουν την αίτηση εγκαίρως. Έχουμε πάρα πολλούς Βρετανούς να ζουν στην Ιταλία και πάρα πολλού νέους. Όχι μόνο θα πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα διαμονής, αλλά πρέπει να αποκαταστήσουμε και την ελπίδα να μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους στην Ιταλία και να οικοδομήσουν εκεί μια νέα ζωή. Αυτό επίσης είναι ένα θεμελιώδε δικαιώμα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ. Πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και του είπε ο Μπόρι Τζόνσον και ο Μάικλ Γκόβορ ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτομάτω αναγνωρίζει το δικαίωμά του στην παραμονή και ε, συνεχίζουν να διατηρούν τα δικαιώματα που είχαν και πριν από το Brexit. Ο Ντάνιελ Άνταμ είπε ότι είναι ε, ανεύθυνο να φοβίζουμε και να τρομάζουμε του ε, πολίτε λέγοντα ότι θα αλλάξει το καθεστώ του μετά το Brexit. Ακόμα και ο Νάτζελ Φάρατζ είπε ότι μπορούν να παραμείνουν και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με του Βρετανού υπηκόου γιατί να υπαναχωρήσουμε σε αυτό ουσιαστικά θα μας έκανε τριτοκοσμική χώρα. Όμως και πάλι τι βλέπουμε εδώ σήμερα. Πολύ γρήγορα αυτή η αυτόματη αναγνώριση έχει ε, ε εξοκύλει σε μια συζήτηση για μη αναγνώριση ακόμα και απέλαση ορισμένων πολιτών. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι πολλοί Πολλέ ευπαθεί ε, κοινωνικέ ομάδε ε, διακινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματά του. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την ε, ανησυχία και αγωνία στον Ηνωμένο Βασίλειο σε του Ευρωπαίου πολίτε, γιατί πολλοί έχουν ζήσει και βιώσει αυτή την απώλεια δικαιωμάτων. Και αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να γίνει μπανανία εντό αγωγικών, μπορεί να το κάνει μετά τον Brexit. Αλλά τα τρία εκατομμύρια πολίτε Ευρωπαίοι πολίτε που μένουν στο, Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπό δική μας ευθύνη και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν τα μεγαλύτερα θύματα του Brexit. Αυτή είναι η θέση, η πάγια θέση του Κοινοβουλίου από την αρχή. Γι' αυτό και τώρα έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε πόσο σοβαρά έχουμε πάρει αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιονγκέριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 31 Ιανουαρίου Βλέπουμε ότι θα φύγει ε, το Νέο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλησιάζει αυτή η ημερομηνία και μέχρι ε, το Ιανουάριο του 2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η συζήτηση. Ελπίζουμε να υπάρχει συμφωνία για τις μελλοντικέ σχέσεις, αλλά εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες, ε, οι εργαζόμενοι που καταβάλουν το μεγαλύτερο τίμημα σε αυτό το διαζύγιο πρέπει να ακολουθήσουμε τα κοινωνικά πρότυπα, να τα υπερασπιστούμε εμείς. Δεν θέλουμε ε, να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αναλάβει τις δεσμεύσεις του σε ό,τι αφορά και τα κοινωνικά επιδόματα και δικαιώματα και απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες ε, που καταβάλουν ε, τα απαραίτητα. Το Brexit δεν αποτελεί ε, καμία δικαιολογία ε, προς μια αρνητική εξέλιξη. Εγώ βέβαια κρατάω την αναπνοή μου. Ο κύριος Κέλεχερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Να πω ότι μιλώ κυρίως ε, στο ε, πλαίσιο ε, της Ιρλανδίας και εκ μέρους των Ιρλανδών πολιτών που ζουν στην Ιρλανδία αλλά και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να δεκτούμε ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ένα συμβιβασμό για τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορούμε να, συμβαστούμε, μάλλον για τα κρατικά προϊόντα, για το εμπόριο, ε, για τις οικονομικές υπηρεσίες. Όμως στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας είναι τα δικαιώματα των πολιτών και θέλω να διασφαλίσω ότι θα τα προστατεύσουμε. Έχουμε κοινό ταξιδιωτικό χώρο με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και κύριε Μπαρνιέ θέλω να διασφαλίσω ότι όταν θα γίνει τρίτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τα δικαιώματα των πολιτών θα διατηρηθούν και θα προστατευτούν. Πολύ απλά πράγματα. Η μη γνώριση των επαγγελματικών προσόντων έχει σημαντικέ επιπτώσει στην Ιρλανδία. Οι άνθρωποι ε, δεν θα μπορούν ε, να εργαστούν σε όλε τι δικαιοδοσίε. Γι' αυτό τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να είναι στη τμήμα αυτή τη συμφωνία ε, και τι μελλοντικέ σχέσει. Δεν μπορούμε να έχουμε συμβιβασμού για τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ένσλι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ως δημοτικό σύμβουλο στο Νότιο Λονδίνο έχω δει το πώς μεταχειρίστηκε την ε, περίπτωση του Windrush ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες από την Καραϊβική που δεν έλαβαν υπηκότητα. Είχαν ζήσει όλη τους τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξαφνικά δεν μπορούν να δουλέψουν, ε, να έχουν παροχές και πρόσβαση στην υπηρεσία υγείας. Παρά την φοβερή αυτή αδικία, η Βρετανική κυβέρνηση προσπαθεί ακριβώς να κάνει τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους να περάσουν από το ίδιο διαλυμένο σύστημα. Ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες ζουν στην περιφερειά μου, στο Λονδίνο. Εγώ είμαι ο Ευρωβουλευτής τους. Δεν θα κάθομαι να κοιτάω ενώ παραβιάζονται τα δικαιώματα τους. Δεν μπορούμε να, υπερασπι... να εμπιστευτούμε αυτήν την Βρετανική κυβέρνηση. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε όλου του ευρωβουλευτέ που θα παραμείνουν σε αυτήν την αίθουσα για τέσσερα χρόνια. Σα παρακαλώ, μην σταματήσετε να μάχεστε για τα δικαιώματα των Βρετανών στις χώρες σας ε, και των υπηκών σας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βοηθήστε μας να λογοδοτήσουν οι κυβερνήσεις μας. Ο κύριος Λιμπεράτσκι για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ε, είπε ο Πρωθυπουργός ο κ. Πλένκοβιτς, ε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Και μας μίλησε το Συμβούλιο, η Κομισιόν, οι πολιτικές ομάδες και βλέπουμε ότι είμαστε ενωμένοι. Οι βασικές μας ανησυχίες είναι οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στο Ενωμένο Βασίλειο, αλλά και οι Βρετανοί που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει και ένα εκατομμύριο Πολωνούς Κάτι το οποίο ανέφερε και η κυρία Φόντερ Λάιεν, ανέφερε τον περίφημο Πολωνό ΣΕΦ, 440 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες επίσης ε, παραμένουν στην Ένωση και, και αυτούς πρέπει να έχουμε κατά νου. Και θα ήθελα να θυμόμαστε και τα 38 εκατομμύρια Πολωνούς πολίτες. Στο διαζύγιο αυτό λοιπόν εμείς είμαστε οι Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το πλέον έκτιμά μας. Ευχαριστώ η κυρία Ίνετφελντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση φυσικά είναι αν οι διευθετήσει θα είναι επαρκείς, αλλά μια άλλη ερώτηση είναι πώ θα εφαρμοστούν. Και εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση Τζόνσον ότι θα το κάνει αυτό ορθά. Και πρέπει να πω ότι τα μηνύματα μέχρι τώρα δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη και ακούω εδώ ότι λέγεται και από τους οπαδούς του Brexit ανησυχώ γιατί δεν είναι και τόσο θερμοί όσο λένε. Και αναρωτιέμαι Ποιο ε, θα ωφεληθεί αν αφαιρέσουμε τα δικαιώματα 5 εκατομμύρια ανθρώπου, Ποιο είναι ο σκοπός 5 εκατομμύρια άνθρωποι να είναι σε ένα λίμπο, γιατί πρέπει να ποινικοποιηθούν, τι έγκλημα διέπραξαν και δεν ε, υπάρχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτή είναι η απάντηση, κανένας δεν ωφελείται. Είναι μια εκστρατεία εκδικητική και ηλίθια κατά ανθρώπων που δεν έχουν κάνει τίποτα λάθο. Καμία δημοκρατία δεν πρέπει να μεταχειρίζεται έτσι του πολίτε. Καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει δικαιώματα από του πολίτε η υπηκότητα είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόβιο, δεν ε, μπορεί να αφαιρείται κατά βούληση. Και γι' αυτό εμείς θα σταθούμε εδώ να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των 5 εκατομμυρίων πολιτών. Ευχαριστώ. Υπάρχει ε, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ρόλαντ. Ένα έτοιμο μπλε κάρτας. Δέχεστε. Όχι. Λυπάμαι κύριε Ρόλαντ. Θα επανέλθω αργότερα. Και η κυρία Γουίντεκομ ε, ζητά να παρέμβει, αλλά ήδη πήρατε το λόγο κυρία Γουίντεκομ. Να περάσουμε στην κυρία Ντάουντινγκ για ένα λεπτό για να βάλουμε σε πλαίσιο τη συζήτηση αυτή. Η τελευταία δημοσκόπηση στον Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων στον Ηνωμένο Βασίλειο προτιμούσαν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 52% έναντι 48%. Το ίδιο περιθώριο που κέρδισε το δημοψήφισμα του Brexit, ε, αλλά έχει αναστραφεί τώρα με πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, χιλιάδες πολίτες μένουν στη δική μου επικράτεια, ε, στην βορειοδυτική Αγγλία και οπωσδήποτε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και ότι οι πολίτες τη χάνουν δικές μεταχείρισεις. Τώρα, κρίσιμα ζητήματα ανακύπτουν για τους πολίτες που έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα εγκατάστασης. Οι δικηγόροι λένε παρά το ότι η κυβέρνηση λέει ότι η διαδικασία θα διαρκεί από μία στους τέσσερις μέρες, κάποιοι ε, μένουν για μήνες χωρίς έγγραφα και δεν μπορούν να εγκιάσουν σπίτι να βρουν δουλειά. Αυτό δεν μας δείχνει ένα σύστημα που σκέφτεται τους πολίτες. Απευθύνουμε έκκληση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουμε ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα τηρήσει τη δεσμεύση της για να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών ε, γιατί ε, μόνο ε, αυτό θα μας οδηγήσει στο να έχουμε και αμοιβαιότητα για τους Βρετανούς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κόρμπετ για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο σωστά συζητάει αυτό το θέμα σήμερα εν ώψη της ψηφοφορίας σε δύο εβδομάδες για την Συμφωνία Αποχώρησης του Βασιλείου. Πολύ σωστά λοιπόν γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί από την αρχή αυτή τη διαδικασία η συντηρητική κυβέρνηση έχει δυσχεράνει πολύ τα πράγματα για του ε, πολίτε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Βασίλειο. Χρησιμοποίησε αυτό το θέμα ω διαπραγματευτικό χαρτί και τώρα δεν δέχεται να του δώσει ένα σύστημα πλήρου εγγύησης. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, η άρνηση τη κυβέρνηση να δώσει ένα τυπωμένο έγγραφο. Αυτό ε, δείχνει ότι ακριβώς ο σχεδιασμός είναι να αποδεικνύει ε, ο πολίτης ε, το δικαίωμά του να παραμείνει στο Βασίλειο απέναντι στον εργοδότη ή στον σπιτονικοκύρη. Είναι αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν του συστήματος. Τώρα βλέπουμε τι κάνει ο Μπόρις Τζόνσον παρότι το 53% ψήφισε υπέρ κομμάτων που ήθελαν νέο δημοψήφισμα. Θα αξιοποιήσει όμω ο Τζόνσον το 43% για να ακολουθήσει πιο σκληρή στάση στο Brexit. Ήδη έχει θεσπίσει νομοσχέδιο για την ε, απόρριψη ε, παραμονή σε πάνω από ένα έτος. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει την μικρότερη δυνατή μεταβατική περίοδο και έτσι θα είναι απολύτω αδύνατο να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα που θα ανακύψουν από τον Brexit. Όμω η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, υπερψηφίσουν τη συμφωνία αποχώρηση και να αξιοποιηθεί η μεταβατική αυτή περίοδο για να εξετάσει αυτό το ζήτημα ε, που έθιξα προηγουμένω. Ούτω ώστε και οι επόμενε γενιέ να χαίρουν των δικαιωμάτων ε, όπως ακριβώς και η δική μας. Έχετε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ρόλαντ, κύριε Κόρμπετ. Να προβλέψω ήδη την απάντησή σας. Όχι, ευχαριστώ. Είναι η απάντηση. Το λόγο για ένα λεπτό η κυρία Νετσίνγκα. Ευχαριστώ. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μπήκε στην ΕΟΚ πριν γεννηθώ εγώ για 47 λεπτά χρόνια, συγγνώμη. Ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες ήξεραν τα δικαιώματά τους ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια φίλη μου που μπήκε και ε, μετακόμισε στο Βασίλειο πριν από 40 χρόνια θεωρούσε ότι ποτέ κανεί δεν απλήξει αυτά τα δικαιώματά της, όμως έχουν αλλάξει αυτά μετά τον Brexit. Η φίλη μου λοιπόν παντρεύτηκε, έκανε τα παιδιά της, ε, πήρε διαζύγιο, εργάστηκε για δεκαετίες και τώρα βρίσκεται κοντά στα 80 και έχει πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων του Brexit στη ζωή της. Όμως υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί άλλοι που ήρθαν στο Νέο Βασίλειο πριν από 40 χρόνια και δεν έχουν ε, τις ίδιες δυνατότητες, έχουν προβλήματα υγείας και θα έπρεπε να κατοχυρώσουμε το δικαίωμά τους στην περίθαλψη, για παράδειγμα. Η τρέχουσα διαδικασία ε, παραμονής δεν είναι εύκολη, ιδίω για αυτούς που δεν έχουν εξοικειωθεί με τέτοιες ε, διαδικτυακές ε, διαδικασίες. Και είναι ακόμα ένα παράδειγμα γιατί ε, δεν εμπιστεύεται ο κόσμος ε, τη συντηρητική κυβέρνηση. Πολλοί έχουν ε, ζητήσει, έχουν κάνει την αίτηση, έχει απορριφθεί. Βρίσκονται λοιπόν σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση που δεν ξέρουν τι μέλη για να είστε και φοβάμαι ότι αυτοί θα τεθούν σε κίνδυνο στο μέλλον. Κυρία Τσόντζ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή μας υπενθυμίζει ότι το Brexit δεν θα γίνει 31 Ιανουαρίου δεν είναι κάτι το απλό όπως λέει ο κύριος ε, Τζόνσον, είναι κάτι το πολύ δύσκολο σαν ένα γεύμα που δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ και θα το μαγειρεύσουν δύο σεφ σε διαφορετικές κουζίνες. Θα μας κάτσει στο, στο μάχη για πολλά χρόνια. Λοιπόν δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, υπάρχουν πραγματικά προβλήματα για το σύστημα αυτό και χρειαζόμαστε περισσότερα, ζητάνε περισσότερα στοιχεία, απειλές, απέλασης ε, κίνδυνος νέου σκανδάλου Windrush σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. είναι μια πικρή ηρωνία το ότι οι ευρωβουλευτές ε, εδώ πέρα έχουν περισσότερο μεγαλύτερο λόγο για το θέμα αυτό από ότι οι Βρετανοί βουλευτές γιατί πλέον δεν έχει άλλο λόγο το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν δεν λειτουργεί Έχουμε πολλά να διαπραγματευτούμε, λίγο χρόνο και υπάρχει κίνδυνος ακόμα να μην υπάρξει συμφωνία. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, εγώ και οι συναδελφοί μου, για να επιδιορθώσουμε την δημοκρατία μας και να ελέγξουμε την κυβέρνησή μας. Σταθείτε παρακαλώ στο πλευρό μας για να υπερασπιστούμε τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες μας και τα δικαιώματα των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Τσάουνς. Ο κύριος Ρόλαντ ε, ζητάει για τρίτη φορά μπλε κάρτα. Δέχεστε. Δεν βλέπω κάποιον λόγο για να ακούσω ακόμη περισσότερο τα πεδαριώδη επιχειρήματα και τις προκαταλήψεις του, Brexit, του κόμματος Brexit. Κύριε Ρόλαντ, μάλλον όχι ήταν αυτό. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γκαρικάνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω το θέμα αυτό του καθεστώτος εγκατάστασης ε, και του τυπωμένου χαρτιού. Έχω πολλούς φίλους, ε, τους έχω επισκεφθεί στο Λονδίνο και αλλού και μου λένε ότι το σύστημα είναι πραγματικά άδικο και δημιουργεί αβεβαιότητα. Το βασικό είναι ότι τους στέλνουν ένα PDF με email, το οποίο μπορούν να τυπώσουν, αλλά μπορεί να το πλαστογραφήσει ο καθένας, που λέει ότι έχουν άδεια παραμονής. Δεν έχουν κάποια κάρτα για όταν ταξιδεύουν, δεν έχουν κάποια κάρτα όταν πάνε στη δουλειά τους, δεν ξέρουν αν την επόμενη φορά που θα μπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν θα του αφήσουν. Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή λύση. Μια κάρτα με τη φωτογραφία τους που μπορούν να έχουν όπως είναι η κάρτα παραμονή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, οι πολίτε μα εδώ πέρα υφίστανται μια αδικία, ένα σύστημα το οποίο είναι άκαρδο και θα πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση με τις ε, Βρετανικές αρχές για να υπάρχει κάτι απτό στα χέρια των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ρίτσι για ένα λεπτό. Το μεγάλο θέμα σήμερα ε, έχει να κάνει με δύο μέρη. Τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα δικαιώματα των Βρετανών ε, στα 27 κράτη-μέλη. Όμως το υποκείμενο πρόβλημα είναι το ίδιο. Ε, έχουμε ακροδεξιό, δικτατορικό, εθνικιστικό λαϊκισμό και ε, βλέπουμε ότι απειλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμεί οι Ευρωπαίοι στη Βρετανία, με νύχια και με δόντια θα αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα ε, και ε, ε, δυστυχώς έχετε εσείς μάλλον συγγνώμη την εξουσία και την αρμοδιότητα να προστατεύσετε τους Βρετανούς πολίτες. Ε, πρέπει να είστε γενναιόδοροι απέναντί μας. Για να παραφράσω το Σοκράτη, δεν είμαι μόνο πολίτης της Σκοτίας και της Βρετανίας εγώ, αλλά της Ευρώπης και του κόσμου. Και δεν θέλω να χάσω κανένα, καμία από αυτές τις ταυτότητες. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρόλαντ, ε, κυρία Ρίτσι, θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε θα παραπέμψω στην απάντηση της ε, προλέλησης σας. Και πάλι υπάρχει άρνηση, λυπάμαι. Να περάσουμε στην κυρία Βονβίζα για ένα λεπτό Ευχαριστώ. Είμαι μία από τα τρία εκατομμύρια πολίτες ε, που τους αρνήθηκαν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα το 2016. Έχω τώρα βρετανικό διαβητήριο, μου κόστησε 15.000 λίρες. Πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν ε, αυτό το ποσό, ακόμη και αν ε, έχουν τις προϋποθέσεις. Βλέπουμε τώρα ότι η βρετανική κυβέρνηση αναπτύσσει μια εχθρική στάση. ζητήσαμε από την κυβέρνηση να μειώσει το τέλος ε, για να γίνει κανείς επίκος. Όμως αυτό είναι το ένα, το να χάσει την επικότητα είναι το άλλο. Θα πρέπει να επιτρέψουν τα κράτη-μέλη στου Βρετανού πολίτε να διατηρήσουν την αρχική του υπηκότητα, είτε γίνουν Βρετανοί κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου, είτε μετά. Είναι ζωτικό να ξέρουν ότι δεν θα χάσουν τα δικαιώματά του ω Ευρωπαίοι πολίτε. Ε, και τέλο, ε, ευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ε, μία υπηκότητα σύνδεση για πολλού πολίτε που θέλουν να παραμείνουν κοντά στου ευρωπαϊκού γείτονε και θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τι ελευθερίε εταιρείε ε, δυνάμει τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι καλό για του ε, πολίτε τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και για του Βρετανού πολίτε, αλλά είναι και καλό για να συνεχιστούν οι φιλικέ σχέσει που επιγόντω χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόλαν θέλει να σας θέσει μια ερώτηση, θα δεχτείτε. It's another no. Και πάλι όχι. Δεν είμαι ναι, προσωπικό, είμαι σίγουρη, αλλά αρνήθηκε η συνάδελφος. Ε, να περάσουμε στο Κατσιδιά, κύριο Σκέλη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είτε μας αρέσει το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε όχι, αυτό το σύστημα έχει. Τώρα λοιπόν ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε την ε, πλειοψηφία, θα ολοκληρωθεί το Brexit εντό λίγων ημερών. Ε, η χώρα μου βέβαια, η Ιρλανδία, θα είναι αυτή που θα λυπηθεί περισσότερο για αυτή την εξέλιξη. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τους ε, κοινούς μας ε, δεσμούς. Ευχαριστώ όλους ε, τους Βρετανούς συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου εδώ και πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν την πραγματικότητα, πρέπει να την αποδεχθούμε και να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Να συνάψουμε μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. Χρειάζεται λοιπόν καλόπιστο πνεύμα από όλες τις πλευρές και όπως είπε και ο κύριος Βρεχόφστατ, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, το ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλιώ δεν πρόκειται να περάσει η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Αυτό είναι το μέλημά μα λοιπόν τώρα, να γίνει σωστά αυτή η διαπραγμάτευση για την Ζώνη Ελευθερών Συναλλαγών. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ward. Εγώ καθώς και εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες και Βρετανοί υπήκοοι σύντομα θα στερηθούμε πολλά μας ε, δικαιώματα εξαιτίας ε, μιας ε, πολύ κακοσχεδιασμένης και κακά ελοποιημένης διαδικασίας ό,τι φορά το Brexit. Έχουμε λοιπόν πολύ δυσάρεστες εξελίξεις που δεν έχουν καμία σχέση με μια δυτική δημοκρατία κατηγορίες που πλήττονται περισσότερο από τον Brexit δεν είχαν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη. Όλοι οι νέοι που θα περιοριστούν οι δυνατότητέ του στο μέλλον ε, τα παιδιά μεταναστών που αρνούνται να εξετάσουν οι ε, συντηρητικοί, τα εκατομμύρια πολιτών που ζουν, μελετούν, εργάζονται, σπουδάζουν και καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Νέο Βασίλειο και πολλές άλλες ε, κοινωνικές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι που αποκλείονται από το σύστημα κοινωνικής ε, προστασίας. Έχουμε, λοιπόν, ε, θα έχουμε μια επανάληψη του σκανδάλου Windrush που είδαμε στο μεγάλο, ε, στο, στο Βασίλειο. Και βλέπουμε ότι ένα κομμάτι κρέας θα έχει περισσότερα δικαιώματα κατά την διάσχεση των συνόρων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Μεγάλης Βρετανίας από ότι ένας άνθρωπος. Αυτό μας κάνει τελικά ένα κομμάτι κρέας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρόλαντ έχει ένα ερώτημα για σας δεν βλέπω κανένα λόγο να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ε, το δικαίωμα να πάρουν τον λόγο εδώ όταν δεν έρχονται στις επιτροπές για να κάνουν τη δουλειά τους. Ας έρθουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να βγάλουν τα λεφτά τους αντί να έρχονται εδώ και να διχάζουν ε, τους ε, βουλευτές. Συγγνώμη, η απάντηση είναι όχι. Η κυρία Κίψον έχει το λόγο. Not now. Ευχαριστώ. Θα πάρω το λόγο ε, για να υπερασπίσω τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, έχουμε πολίτε που χάνουν σημαντικά δικαιώματα τα οποία κατήχαν ε, για δεκαετίε. Έγιναν υποσχέσει, σαν οι άνθρωποι το σπίτι του, μετακόμισαν, άλλαξε τη ζωή του, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, έκαναν σχέδια για το μέλλον. Και τώρα λόγω κάποιων πολιτικών και ενό πολιτικού συστήματος που δεν λειτουργεί, δεν γίνονται σεβαστές υποσχέσει. Ε, τώρα, οι πολίτες ε, που εργάζονται, ζουν και πληρώνουν φορού, ε, τους αντιμετωπίζουμε ως εξωγενείς. Και τι γινόταν ε, ε, εδώ και πολλά χρόνια όταν δεν ε, χρειαζόταν υποτίθεται να έχουν αυτά τα έγγραφα. Ζούμε σε βεβαιότητα. Αυτό μας είναι λάθος. Αυτό το κοινοβούλιο είναι σε θέση να στείλει ένα λάθητο μήνυμα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Παρακαλώ στείλτε το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπρουτζίνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπαρνιέ στις συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και με τη Βρετανική κυβέρνηση να μην παρασυρθεί από αυτά τα συναισθήματα που βλέπουμε να κυριαρχούν και στα δεξιά και στα αριστερά αυτού του ημικυκλίου. Αυτή η συμφωνία αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνταχθεί και λόγω όλων αυτών των συναισθημάτων δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η τύχη όλων αυτών των πολιτών μεταξύ αυτών ε, και πολλοί Πολωνοί ε, οι οποίοι έχτισαν κατά κάποιο τρόπο ε, την Βρετανική οικονομία. Εγώ άκουσα με πολλές φορές Βρετανούς να μιλούν για Πολωνούς και μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν μόνο Πολωνοί σεφ και αστυνομικοί παραδείγματος χάρη και Κάποιοι Πολωνοί έλεγαν ότι θα ήθελαν να μπορούν να επιστρέψουν στην Πολωνία, όμως έλεγαν ότι είχαν φτιάξει την ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλοί θέλουν να μείνουν. Πρέπει λοιπόν να μην παρασυρώμαστε από τα συναισθήματα, αλλά να είμαστε λογικοί. Και να πω ότι ε, υποτίθεται ότι ο Χάρη και η Μέγκαν ε, έχουν διαλέξει ε, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Κύριο Φερέιρα, θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα δίκαια των πολιτών που ζουν και εργάζονται στο Ρωμένο Βασίλειο αλλά και όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο των σημερινών αλλά και αυτών που στο μέλλον σχεδιάζουν κάτι τέτοιο τέτοιο. Ε, δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκή στο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών. Ας ε, θυμηθούμε τι υπόθηκε στον ε, κύριο Κάμερον για το δημοψήφισμα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε τι ασφαλιστικέ δικλείδε για τα δικαιώματα των εργαζομένων και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα παραμονή μη διαχειριστική μεταχείριση, πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, τη φορητότητα των δικαιωμάτων, την κοινωνική ασφάλεια εις ε, την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα. Και ε, συζήτηση που θα συνεχιστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τα περιλαμβάνει αυτά, αλλά και στις διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ κάθε κράτου μέλους και του Ηνωμένου Βασίλειου για να έχουμε μελλοντικέ διμερείς ε, σχέσει που θα του ωφελούν όλου. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πέντε ομιλητέ στο ΚΑΤΣΔΙΑΕ και θα δώσω τώρα το λόγο στο Μισελ Μπαρνιέ για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, του ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, ε, πάντα σας